τον, ε, ε, την 5η 17 Απριλίου. Αύριο θα ξεκινήσει η Διεθνής ξεκινησει η διεθνη ημερα που είναι αφιερωμένη στις τα τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορίας. Είναι αφιερωμένη στις γυναίκες και ε, στόχο έχει να προωθήσει την ενασχόληση των γυναικών με τους τομείς της πληροφορικής, της μηχανικής και των μαθηματικών, ενώ τομέα που είναι σε διεύρυνση. Στην Ευρώπη 75.000 ε, ε, ε, γυναίκες έχουν πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης έναντι 95.000 ανδρών ετησίως. Δυστυχώς πολύ μικρό ποσοστό εξ αυτών βρίσκουν εργασία σε αυτό το τομέα. Οι γυναίκες καλύπτουν το 24% των θέσεων απασχόλησης στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα και κυρίως σε διοικητικές θέσεις, για διοικητικές θέσεις πρόκειται και το χάσμα των μεταξύ των δύο φύλων μεγαλώνει όσο ανεβαίνουν στην ιεραρχία. Ανεβαίνουμε στην ιεραρχία. Επίσης, ε, ο γυναικείος πληθυσμός που έχει πρόσβαση στο ίντερνετ είναι πολύ μικρότερος, κατά 12% του ανδρικού πληθυσμού και αυτό το ποσοστό δυστυχώς έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Εύχομαι η αυριανή ημέρα να χρησιμεύσει ως λαβή για έμπνευση, για να εργαστούμε μαζί, για να εγγυηθούμε στις νέες όλου του κόσμου ένα καλύτερο μέλλον. Θα πρέπει αυτός να είναι ένας στόχος ε, μεταξύ των στόχων ε, για την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ μεταξύ των δύο φίλων που και στον τομέα της επικοινωνίας ε, και της πληροφορικής. Θα πρέπει λοιπόν τα συστήματα παιδείας μας να είναι για καθολικά και να ενθαρρύνουν τις νέες εταιρείε να άρουν τους φραγμούς των φίλων και να θαρρύνουν τις γυναίκες εργαζόμενες. Καλή εργασία.